Uh, welcome to everybody. We can start now. Yesterday we had a very, very intense... Καλημέρα σας ε, κυρίες και κύριοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε νομίζω. Χθε είχαμε κατάμεστο πρόγραμμα. Εργαστήκαμε άοκνα. Ελπίζω να έρθουν και άλλοι συνάδελφοι στο μεταξύ, αλλά θέλω να είμαστε ευγενείς και απέναντι στους καλεσμένους μας. Περνάστε τελικά. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να ξεκινήσουμε σήμερα με ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θέλουμε να το εμβαθύνουμε περισσότερο σχετικά με τα πεδία με τα οποία καλύπτουμε σαν Επιτροπή. Γνωρίζετε ότι σαν Επιτροπή Πολιτισμού και σαν Κοινοβούλιο θεωρήσαμε ότι παράλληλα με τις προτεραιότητες που καθορίζονται στα πλαίσια του στρατηγικού προγράμματος ε, της Επιτροπής να συμπεριληφθούν ε, και οι λεγόμενες ε, βιομηχανικές δραστηριότητες στον τομέα της πνευματικής δημιουργίας και η εκπαίδευση. Και θέλουμε να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε σήμερα στα διάφορα κράτη-μέλη γύρω από αυτό. Να καλωσορίσω τον Χάραλ Γκρούμπερ, ο οποίος είναι υπεύθυνο για τέτοιου είδους θέματα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να πω επίσης ότι στις 3 Δεκεμβρίου στην διακυβερνητική η οποία είχε σαν βασικό θέμα την εκπαίδευση και την νεότητα και που οργανώσαμε στις Βρυξέλλες, ο κύριος Γκρούμπερ ήταν ένας επιμελής ε, συμμετέχων στις εργασίες. Δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο και παρόλα αυτά πήρε και αυτός μέρος και προσέφερε και αυτό στην δική του συνεισφορά και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είπε ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να επενδύσει στις υποδομές της εκπαιδευτικής αλλά και στην ψηφιακή ε, παραγωγή. Υπάρχει μια ανηλυμένη υποχρέωση της ε, ΜΠΕΗ εδώ και χρόνια για την απασχόληση των νέων ένα πρόγραμμα που προσφέρει ειδικέ ε, δανειοδοτήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να απασχολούν νέους και να παρέχουν και μια επαγγελματική κατάρτιση προς αυτούς. Θα έλεγα ότι θα δώσουμε αμέσω το λόγο στον κύριο Γκρούμπερ για να μας μιλήσει επί της ουσίας. Γνωρίζουμε ότι το πρόγραμμα επενδύσεων που έχει ανακοινωθεί, το λεγόμενο πρόγραμμα Juncker, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει και μέσω αυτών των νέων τρόπων εγγυήσεων που παρέχει να επιτρέψει και στους ευρωπαϊκούς εταίρους και στους ευρωπαίους εταίρους συγγνώμη και στις, στους εθνικούς εταίρους την δυνατότητα να επενδύουν σε τομείς στους οποίους ε, ο κίνδυνος εισαγωγικά για τις επιχειρήσεις είναι αρκετά υψηλός. Και έτσι λοιπόν να δίδονται περαιτέρω εγγυήσει σε τομείς όπου η απόσβεση θα έλεγα, η απόδοση δεν είναι άμεση, προϋποθέτει όμως μια εμπειρογνωμοσύνη ε, τέτοια η οποία θα οδηγήσει στην απόσβεση μέσω πρόθεσμα αλλά θα, ε, αυτού του είδους η επένδυση θα είναι ευρύτατη σημασίας και θα παίξει συνεκτικό κοινωνικά ρόλο. Είναι λοιπόν περίπλοκο το θέμα και γι' αυτό η στρατηγική αυτή την οποία, ε, στην οποία στοχεύουμε θέλουμε να είναι σωστά προσανατολισμένη. Υπήρξε πρόσφατα μια συμφωνία ανάμεσα στην Προεδρία του Κοινοβουλίου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και την υπηρεσία εκδόσεων έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στους πιθανούς επενδυτές στις διάφορες χώρες σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις εθνικές υπηρεσίες να δείξουμε σε αυτούς οι οποίοι έχουν την δυνατότητα επένδυσης και δεν το κάνουν τι τι πεδίο θα έλεγα πιθανό επενδυτικό είναι ανοιχτό μπροστά τους. Έτσι θα υπάρξουν κάποια συγκεκριμένα προγράμματα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εκπροσωπείται άλλωστε σήμερα και από τις δύο γενικές διευθύνσεις αλλά βρισκόμαστε τώρα στην προκαταρκτική φάση και ο κύριος Γκρούμπερ θα μας παρουσιάσει ακριβώς τη σημασία αυτών των συμφωνιών και θα μας παρουσιάσει επίσης και την ιστο, ε, σε εισαγωγικά θύρα την οποία θέλει να δημιουργηθεί ε, γύρω στα 10 λεπτά εν πάση περιπτώσει έχετε το λόγο και μετά θα πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ κυρία Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Παρουσίασα ορισμένες διαφάνειες Illustrate to you what the bank is doing in the domain. για να εξηγήσω το τι κάνει η τράπεζα στα πλαίσια της ανεργίας των νέων, της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων. Θα ήθελα να εκφράσω και κάποιες σκέψεις επίσης για συγκεκριμένους τομείς οι οποίοι αφορούν τη δική σας επιτροπή. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή είναι μία εικόνα των δραστηριοτήτων μας του προηγούμενου έτους. Αυτή είναι η βασική στόχη της πολιτικής της τράπεζάς μας για την ανεργία των νέων ή για την απασχόληση καλύτερα των νέων σε δύο βασικά τομείς ο ένας είναι ο τομέας της καινοτομίας, εδώ είναι θέμα εκπαίδευσης δηλαδή, θεωρούμε ότι η εκπαίδευση είναι μια δυνατότητα η οποία θα καταστήσει ικανούς τους εταίρους να καταστήσουν και αυτοί με τη σειρά τους ανταγωνιστική την οικονομία. Και το δεύτερο στρώμα δραστηριοτήτων είναι οι μικρομεσαίες. Οι μικρομεσαίες είναι αυτές οι οποίες στην ουσία ε, δίνουν την δυνατότητα απασχόλησης στους νέους, δημιουργούν θέσεις απασχόλησης για τους νέους. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία όταν αναφέρεται κανείς στην τράπεζά μας είναι ότι χρηματοδοτεί συγκεκριμένα σχέδια επενδυτικά και προγράμματα. Ο βασικός στόχος είναι να δίνουμε δάνεια αλλά τα δάνεια αυτά θα πρέπει να στηρίζονται, να βασίζονται σε ένα σχέδιο, σε ένα πρόγραμμα. Πρέπει να είναι συγκεκριμένα και προσδιορισμένα. Ήδη το ίδιο το σχέδιο, το πρόγραμμα αποτελεί ένα αγαθό. Μπορεί να είναι κάτι το απτό, δηλαδή υποδομή οδική, τηλεπικοινωνική ή και μη απτό, δηλαδή έρευνα και ανάπτυξη γενικότερα. Είναι ένα αγαθό γνωστικό, ε, χωρίς αμφιβολία λοιπόν είναι ένα συγκεκριμένο αγαθό γιατί δημιουργεί προϋποθέσεις για μελλοντικά κέρδη και εισοδήματα. Για τη νεότητα. Η νεότητα είναι ακριβώς το μεγάλο πλεονέκτημα της Ευρώπης και δεν το χρησιμοποιούμε σοφά, δεν επενδύουμε επαρκώς η τράπεζα λοιπόν αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επενδύσουμε στους νέους σαν ένα πολύτιμο αγαθό. Πρέπει να προωθήσουμε τις δυνατότητες και τις ικανότητες των νέων για να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους, γιατί τότε θα έχουμε χαμένες γένειες, χαμένα έσοδα, χαμένο πλούτο. Είναι βασική ανησυχία για την τράπεζά μας δηλαδή αυτό. Είναι δημιουργία δηλαδή περαιτέρω αγαθών. Η τράπεζα βέβαια δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει προγράμματα τα οποία δεν είναι καλά τεκμηριωμένα και υπάρχουν συγκεκριμένοι παράμετροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ποιότητας ενός προγράμματος. Είναι κάτι που έχει κοινωνικό όφελος, είναι κάτι το οποίο είναι τεχνικά βιώσιμο, είναι οικονομικά δικαιολογημένο, και μπορεί να αυτοχρηματοδοτηθεί, είναι βιώσιμο δηλαδή χρηματοδοτικά. Ε, το πρόγραμμα αυτό με λίγα λόγια είναι ικανό να βρει τις ε, επαρκείς μορφές χρηματοδότησης για να επιστρέψει το δάνειο το οποίο έχει πάρει. Αυτές είναι οι βασικές ανησυχίες της τράπεζας όταν έχουμε να κάνουμε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ε, σχετικά με το πρόγραμμα για τη βελτίωση των ικανοτήτων και την επένδυση στην κατάρτιση των νέων. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προχώρησε με μεγάλη ταχύτητα. Ήδη από το 2013 έγιναν οι αρχικές προτάσεις οι οποίες έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο. Θα σας πω κάποιες λεπτομέρειες εδώ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν επίγον και γι' αυτό προχώρησε πολύ γρήγορα η τράπεζα ξεκίνησε με ένα βραχυπρόθεσμο λοιπόν πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. έξι δις κατέτος σε δύο βασικά πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι οι επαγγελματικές ικανότητες. Δηλαδή η πλευρά της προσφοράς προς την αγορά εργασίας. Υπάρχει ανάγκη να δώσουμε στους νέους τις επαρκείς ικανότητες να προσαρμόσουν ε, την προσφορά τους προς την αγορά εργασίας. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Τρία δις σε αυτό το σκέλος και στο άλλο είναι η ζήτηση. Ποιος προσλαμβάνει τους νέους, βασικά οι μικρομεσές. Δίδουμε κίνητρα λοιπόν στις μικρομεσές έτσι ώστε να προσλάβουν... Uh, Νέο προσωπικό. Στην πλευρά της ζήτησης υπάρχουν κάποια μέσα τα οποία ήδη προπήρχαν και ενισχύθηκαν. Υπάρχει το θέμα της ε, μικροχρηματοδότησης ε, και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όπως επίσης και οι ε, εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης που μεσολαβούν μερικές φορές στα πλαίσια της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων. Δεν έχουμε λοιπόν τώρα χρόνο για να περάσουμε σε λεπτομέρειες γιατί όλα αυτά έχουν γίνει σε μικρό χρονικό διάστημα. Πρέπει να ξεκινήσουμε ήδη από τον επόμενο μήνα και έπρεπε να ξεκινήσουμε μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και το πρόγραμμα αυτό συνεχίζει να εξελίσσεται. Τώρα, στον τομέα της απόκτησης περαιτέρω ικανοτήτων. Εν πολλής ε, τα θέματα έχουν σχέση εδώ με τις υποδομές. Ε, υπάρχει έλλειψη επενδύσεων στις υποδομές τις εκπαιδευτικές ο προϋπολογισμός ε, για την εκπαίδευση σύμφωνα με τα δεδομένα του ΟΣΑ θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένα το 10% συνολικά. Ε, το, αλλά στις περισσότερες χώρες είναι πολύ λιγότερο. Ε, μπορεί βέβαια να λειτουργεί ένα σχολείο ακόμα και αν μισογκρεμίζεται θα έλεγε κανείς και να το καθυστερεί αλλά παρόλα αυτά ε, η προσπάθεια είναι να μην θυγούν τα δημοσιονομικά. Και αυτό που κατανοήσαμε είναι ότι στον τομέα των υποδομών ε, είναι κάτι το οποίο είναι μια μακροπρόθεσμη συγκεκριμένη επένδυση και εκεί εμείς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, εκεί μπορούμε να είμαστε παραγωγικοί. Ε, διευκολύνουμε λοιπόν τις επενδύσεις στις υποδομές κάτι το οποίο σε επίπεδο ποιότητας επιτρέπει τη σωστότερη παροχή υπηρεσιών στους εκπαιδευομένους και βρίσκεται η εκπαιδευτική μονάδα στον σωστό χώρο γιατί πολλές φορές κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Όλες αυτές είναι ανησυχίες οι οποίες την τελευταία δεκαετία αγνοήθηκαν. Και δεύτερον προσπαθούμε να βελτιώσουμε και κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι μη ε, θα έλεγα υλικές χρησιμοποιούμε σαν αγαθά τα προγράμματα αυτά, ε, τα σχολεία. Προσπαθούμε δηλαδή σαν τράπεζα να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε επιμέρους εκπαιδευτικά προγράμματα από συγκεκριμένες μονάδες εκπαίδευσης, πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τους εκπαιδευτές όχι μόνο δηλαδή προγράμματα για τους εκπαιδευομένους αλλά και για τους εκπαιδευτές έτσι ώστε να είναι θα έλεγα επίκαιρη η γνώση τους σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ταυτόχρονα να διευκολύνουμε επίσης μέσα για την εκπαίδευση όπως τα φοιτητικά δάνεια, η κινητικότητα, η σπουδαστική, όλα αυτά είναι τομείς στους οποίους διευκολύνουμε τη χρηματοδότηση. Είναι άνηση βέβαια η κατανομή. Η καθημερινότητά μας βασικά είναι οι υποδομές, είναι οι κτηριακές υποδομές, τα δίκτυα κτλ. Ε, στο φάκελο υπάρχουν πολλά παραδείγματα, δείχνουμε πως τέτοιου είδους επενδύσεις μπορεί να πραγματοθούν. Υπάρχει ακόμα πολύ περαιτέρω θα έλεγα δυνατότητα παρέμβασης στον τομέα του λογισμικού ε, για ε, την παρέμβαση και ενίσχυση προγραμμάτων από την τράπεζα. Λοιπόν, βλέπετε εδώ μια συγκεκριμένη αναφορά των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων μας για τον προηγούμενα χρόνια. Βλέπετε ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους είχαμε θέσει και τους οποίους ξεπεράσαμε. Ήδη από πέρυσι υπήρξαν σημαντικές επενδύσεις ε, στον τομέα ε, της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων που οδήγησε σε προσλήψεις. Ε, βοηθήσαμε την εκπαίδευση επίσης των νέων με μεγάλη επιτυχία αλλά και σε επίπεδο ικανοτήτων και γνώσεων που αφορά την τομέα της προσφοράς ε, νομίζω ότι πήγαμε πολύ καλά έτσι δείχνουν τα αποτελέσματα. Εδώ βλέπετε τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε χώρες 2013-2014 υπήρξαν αλλαγές από τη μία χρονιά στην άλλη είναι συγκυριακές λίγο οι αλλαγές γιατί υπάρχουν κάποια μεγάλα προγράμματα ετήσιας διάρκειας κάποια άλλα διετούς αλλά βλέπετε ότι αυτά τα πράγματα από τον ένα χρόνο στον άλλο αλλάζουν παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες δείχνουν τη δραστηριότητα των χωρών που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Δεν υπάρχει κανένα όριο εδώ. Έχουμε βέβαια ένα ελάχιστο πακέτο, αλλά προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο. Μπορείτε να τα δείτε αυτά προσεκτικά στο φάκελο που έχετε μπροστά σας και να περάσω στο επόμενο βήμα. Τι ε, περιμένουμε τώρα με το πρόγραμμα στρατηγικών επενδύσεων. Αυτό είναι κάτι που είδατε επανειλημμένα και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι το πρόγραμμα αυτό εν πολλής δεν αλλάζει τις δραστηριότητες της τράπεζας σε επίπεδο μεθοδολογικό. Η τράπεζα θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί όμως προγράμματα τα οποία θα πρέπει όπως είπα στην αρχή να είναι καλά, να είναι ποιοτικά. Σας είπα ποιοι είναι οι παράμετροι υπολογισμού της ποιότητας, δηλαδή κοινωνική χρησιμότητα, οικονομική βιωσιμότητα και τεχνική εφικτότητα. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια. Υπάρχουν επίσης δύο περαιτέρω διαστάσεις οι οποίες ε, λαμβάνονται υπόψη από την ΕΦΣΗ. Καταρχάς το μέγεθος της, των δυνατοτήτων μας. Η τράπεζα πρέπει να κάνει περισσότερα, να έχει περισσότερα χρήματα και ταυτόχρονα η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει στην ανάληψη ε, μεγαλύτερου επίπεδου κινδύνων. Δηλαδή όχι πάρα πολύ, χωρίς υπερβολές, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να αναλάβουμε περισσότερους κινδύνους από ό,τι στο παρελθόν. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι καθοριστική αυτή η αλλαγή. Η βασική ιδέα είναι ότι ε, θα πρέπει να κινητοποιήσουμε μέσω του προγράμματος στρατηγικών επενδύσεων τα ιδιωτικά κεφάλαια, τις ιδιωτικές επενδύσεις. Ένας τομέας όπως η εκπαίδευση που είναι ένας από τους στρατηγικούς τομείς ε, και σε επίπεδο μεσαίας κεφαλαιοποίησης βλέπετε ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα κριτήρια επιλεξιμότητας έτσι ώστε να γίνει η πραγματικότητα η επένδυση. Αυτό το οποίο ίσως είναι δύσκολο στον τομέα της εκπαίδευσης είναι ότι κατά κάποιο τρόπο είναι ένας τομέας που κυριαρχείται από τις δημόσιες επενδύσεις ο δημόσιος τομέας για μια τράπεζα είναι θα έλεγα ένας καλός οικονομικός εταίρος, δεν δημιουργεί τεράστιους κινδύνους. Από την άλλη είναι πάρα πολύ δύσκολο να κινητοποιήσει ο τομέας από μόνος του ιδιωτικές επενδύσεις για δημόσιου ενδιαφέροντος θα έλεγα προγράμματα. Το θέμα είναι πώς να κινητοποιήσουμε λοιπόν ιδιωτικές επενδύσεις Σαν παράδειγμα, οι εταιρικέ σχέσεις θέμενη αξίας είναι ένα από τα προγράμματά μας. Πρέπει να είναι οικονομικά εποφελή φυσικά τα προγράμματα αυτά και θετικά για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ε, επίσης και για άλλους τομείς ε, κινητοποίησης της νεότητας βλέπετε ότι ο ιδιωτικός τομέας παρεμβαίνει ιδιαίτερα σε τομείς όπως η επαγγελματική κατάρτιση. Υπάρχουν τομείς όπου ο ιδιωτικός τομέας είναι ιδιαίτερα ικανός για την διδασκαλία των νέων σχετικά με τις ε, απαιτήσει ε, των γνώσεων και των ικανοτήτων τους. Θέλουμε λοιπόν εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία να προωθούνται από επιχειρήσεις γιατί για την επιχείρηση η εκπαίδευση είναι ένα επιπλέον κόστος η εξήγηση του όταν κάποιος στέλνει κάποιον στο σχολείο από μια επιχείρηση. Επίσης ή όταν αποστέλλεται σε μια επιχείρηση να εκπαιδευτεί είναι κάτι το πάρα πολύ ε, σημαντικό σε επίπεδο κατάρτισης. Αναπτύσσονται κοινωνικές ικανότητες και δυνατότητες και ε, δυνατότητες εργασιακές. Οι επενδύσεις λοιπόν υπάρχουν εδώ από πλευρά των επιχειρήσεων. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε αυτού του είδους τις δαπάνες σαν επενδύσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις και τα οποία μπορεί να υποστηριχθούν με διάφορους τρόπους από τη δική μας χρηματοδοτική παρέμβαση. Εδώ βλέπουμε ένα γράφημα το οποίο δείχνει κατά κάποιο τρόπο ε, την ποικιλία των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της τράπεζας ε, και στα πλαίσια του ΕΦΣΥ, του στρατηγικού προγράμματος Juncker από πολύ μικρά προγράμματα μέχρι πάρα πολύ μεγάλα προγράμματα. Επαγγελματική κατάρτιση προωθείται από τον ιδιωτικό τομέα, υψηλού κινδύνου επίσης. Πρέπει να, θα έλεγα, να μπαίνουν σε ένα ευρύτερο σύνολο σε διαφορετικούς, από διαφορετικούς τομείς όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή όταν είναι θα έλεγα υψηλής, μεγάλης ποσότητας τα προγράμματα αυτά ε, τότε μπορεί να μπαίνουν σε ένα ευρύτερο σύνολο από την ίδια την τράπεζα. Τώρα οι εταιρικές σχέσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα PPP, πρέπει να δούμε ποιοι είναι κάποιοι τομείς στους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε είναι η πνευματική δημιουργία. Εδώ σαν παράδειγμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες βοήθειας προς μικρομεσές, προς συνεταιριστικές συνεργατικές οργανώσεις Όλα αυτά μπορούν να, ε, ε, ε, υποστηριχθούν και στα πλαίσια του στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της τράπεζάς μας. Υπάρχει λοιπόν σαφώς εδώ μια δυνατότητα εμπλοκής και με ιδιωτικά προωθούμενες δραστηριότητες. Ε, συνεισφέρουμε όλοι μαζί έτσι στους στόχους του FC, του επενδυτικού προγράμματος. Απαιτείται δημιουργική σκέψη για τον τρόπο πρότασης των προγραμμάτων αυτών. Ε, το πρόγραμμα το επενδυτικό έχει δημιουργήσει ένα κέντρο συμβουλευτικό, ένα advisory hub το οποίο δίδει τους σωστούς προσανατολισμούς έτσι ώστε να βρεθούν τα προγράμματα τα οποία είναι πιθανό να μπορούν να, επενδυτι να βοηθηθούν από τις διαφορετικές επενδυτικές μας δραστηριότητες. Υπάρχει δηλαδή ένα αρκετά ευρύ πεδίο έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρέμβουμε. Απαιτείται όμως προσεκτική δουλειά, απαιτείται δημιουργική σκέψη και από πλευράς των κοινοτήτων που αναζητούν την χρηματοδότηση. Δεν είναι πρόβλημα η χρηματοδότηση. Το θέμα είναι ότι έχουμε στενοπού στη δημιουργία των, προγραμμάτων που να είναι επιλέξιμα για να υποστηριχθούν από τα χρηματοδοτικά μέσα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Γιατί εκεί όλα δεν υπάρχουν. Οπότε αν υπάρχουν ωραία προγράμματα στις ε, δημιουργικές, στους δημιουργικούς κλάδους και στον εκπαιδευτικό τομέα δεν υπάρχουν όρια. Από τη στιγμή που κριθούν επιλέξιμα μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Δεν είναι πρόβλημα η χρηματοδότηση, αλλά θα πρέπει να είναι σωστά σχεδιασμένα, η σύλληψή τους να είναι κατάλληλη. Έχω και μερικά παραδείγματα. Δεν ξέρω τι προτιμάτε. Μπορώ να σας δώσω και κάποια παραδείγματα ή αν προτιμάτε να βάλω τελεία εδώ. ma anche le industrie culturali e creative ci capire. μικροφώνου η πρόεδρος δεν την ακούμε. Είπατε κάτι για τα θέματα της εκπαίδευσης, αλλά για τις ε, βιομηχανίες που έχουν κάποια δημιουργικότητα, πώς προτείνετε να ενθαρρύνουμε κάποια δίκτυα που δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στον τομέα αυτό των κλάδων που δείχνουν κάποια δημιουργικότητα. Το πρώτο παράδειγμα που έχω εδώ είναι καλό παράδειγμα γιατί αφορά αυτούς τους κλάδους, ε, τους ευρηματικούς δημιουργικούς. Πρόκειται για μια ισπανική τράπεζα που προσπαθεί να προαγάγει ε, κάποια προγράμματα και σχέδια στην ανώτατη εκπαίδευση και χορηγεί φοιτητικά δάνεια ώστε να μπορέσουν οι φοιτητέ να χρηματοδοτήσουν τις σπουδέ τους. Τέτοιου είδους φοιτητικά δάνεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς, όχι μόνο για φοιτητέ. Όταν έχουμε συγκέντρωση σχετικά μικρών δανείων, τα συγκεντρώνουμε, οπότε ε, η αποπλήρωση να συναρτάται από την επιτυχία. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο φοιτητή ε, δεν ε, βρίσκει μια δουλειά και δεν μπορεί να αποπληρώσει, τότε διαγράφεται το δάνειό του. Αλλά πολλοί απασχολούνται, πολλοί φοιτητέ, οπότε μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά του, τα φοιτητικά. Τέτοιου είδου προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τώρα, για τον πολιτιστικό τομέα, στο απτικοακουστικά, χρηματοδότηση ταινιών, μπορούμε να έχουμε τέτοιες δραστηριότητες. Και αν έχουμε αρκετά μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων και μπορούμε να τους ε, συγκεντρώσουμε, να τις συγκεντρώσουμε, μπορούμε να τις στηρίξουμε με χρηματοδοτικονομικά μέσα, όπως τα δάνεια, για παράδειγμα. Σκεφτείτε το. Άλλο παράδειγμα. Υποδομές, υποδομές στην παιδεία. ε, σχολεία που παρέχουν κατάρτιση επαγγελματική. Στη Γαλλία έχουμε ένα παράδειγμα και κάποιες χρηματοδοτικές δυσκολίες εκεί. Αλλά αφιπνίστηκαν οι θύνοντες και αντιλήφθηκαν την επιτακτική ανάγκη χρηματοδότηση και τέτοιων προγραμμάτων. Επίσης, για υποδομές στον πολιτιστικό κλάδο. Θα πρέπει να διαρωτηθούμε αν έχουμε υποδομές που μπορούν να τροφοδοτήσουν τέτοιες δραστηριότητες. Γιατί αν δεν μπορούμε να στηρίξουμε τις δραστηριότητες, τουλάχιστον να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για να αναπτυχθούν, για να προαχθούν με αποτελεσματικό τρόπο. Πολύ συχνά αρκεί μια πλατφόρμα, μια πραγματική που μπορεί να είναι είτε πραγματική είτε εικονική στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, ε, μια τράπεζα χρηματοδότησε, στήριξε πολλά προγράμματα στα ψηφιακά οπτικοακουστικά μέσα. Ε, το ορόβιο, το Angry Birds. Πολύ δημιουργική κλάδη στον τομέα των λογισμικών που ε, σχεδιάζουν τέτοια ψηφιακά παιχνίδια. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες ψηφιακού περιεχομένου που παράγονται στο, στις Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά και στην ε, Ευρώπη έχουμε ταλέντα και ευρηματικούς ε, ανθρώπους. Να μην χρειάζεται να φύγουν στις Ηνωμένε Πολιτείες, να στηρίξουμε δραστηριότητες για να μπορέσουν τα ταλέντα μας ε, να ξετυλίξουν τις ικανότητες τους και στην Ευρώπη, να μην χρειάζεται να φεύγουν στις Ηνωμένε Πολιτείες. Σας ευχαριστώ. Καταλαβαίνουμε ότι το θέμα είναι περίπλοκο Υπάρχει επίσης και το κριτήριο της προσθετικότητας το οποίο πρέπει να λειτουργεί μέσω του στρατηγικού προγράμματος σε σχέση με τα υπόλοιπα. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Κάμερ, Εβερτ και μετά Τρόπελ. Σας ευχαριστώ. Μία ερώτηση έχω που αφορά την παιδεία. Πολύ ευαίσθητος τομέας όπως ξέρετε η παιδεία. Ως προς το περιεχόμενο αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Όταν όμως μιλούμε για ιδιωτικές επενδύσεις Λογικό είναι να περιμένουμε μία απόσβηση και ένα κέρδος, μία αποδοτικότητα των επενδύσεων. Στα εκπαιδευτικά ζητήματα όμως πρέπει να είμαστε πιο συνετοί, γιατί σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκουμε την ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Όταν έχουμε λοιπόν εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικά σχέδια, πώς εξασφαλίζεται τη συμβατότητά τους ε, με τα εθνικά ή περιφερειακά εκπαιδευτικά συστήματα και τις εθνικές ή περιφερειακές αρμοδιότητες. Σε ό,τι φορά την επαγγελματική κατάρτιση ή την ε, επαγγελματική επιμόρφωση, εκεί τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Γιατί οι επιχειρήσεις ε, αναζητούν στην αγορά εργασίας ειδικευμένους εργαζόμενους. Και εκεί Όντως, ε, ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμμετέχει αναλαμβάνοντας κάποιες ευθύνες είτε σε ένα διπλό σύστημα με συμπράξεις είτε προσφέροντας ε, επαγγελματική κατάρτιση. Και αυτό ισχύει και για την επιμόρφωση των νέων, αλλά και για τη διαβίου κατάρτιση των ενηλίκων. Ελπίζω να μην χρηματοδοτούμε μόνο ε, προγράμματα προσοδοφόρα που αποφέρουν ε, οικονομικά μονοφέλη. Αλλά να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα που θα προωθούν την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση. κυρία Τρίπελ, σας ευχαριστώ. Πιστεύετε ότι με τις νέες δυνατότητες που δίνει το ΕΦΣΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, θα μπορέσουν και οι κλάδοι της δημιουργίας ε, να ενημερωθούν επαρκώς και να γνωρίζουν τις δυνατότητες που υπάρχουν. Μπορείτε να μας κάνετε μια επισκόπηση του αριθμού των αιτήσεων που έχετε λάβει και πόσες έχουν γίνει δεκτές για χρηματοδότηση. Επίσης, ποια θα είναι τα νέα μέσα χρηματοδότησης ε, για το κλάδους της δημιουργίας ε, από το πρόγραμμα Creative Europe, Δημιουργική Ευρώπη. Ε, θα θέλαμε και προγράμματα πολιτισμικά μικρής εμβέλειας να ε, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν έτσι για χρηματοδότηση και να διαφυλαχθεί ένα μερίδιο και για αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και το έγγραφο που μας δώσατε. Έχω μια ερώτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, συνήθως ε, δεν έχουν αρκετό προσωπικό για να υποβάλουν τις αιτήσει τους. Ε, ε, το ίδιο και τα holdings, οι όμιλοι. που όμως ε, ιδιαίτεροι μεγάλοι όμιλοι έχουν τέτοια επιμελητική υποστήριξη και ακριβώς έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να υποβάλουν πλήρη προγράμματα και να λάβουν ε, χρηματοδότηση, ενώ αντίθετα οι μικρομεσαίες επιχειρήσει είναι η ψυχή της βιομηχανίας, ιδιαίτερα στην Γαλλία. Θα πρέπει να υποστηριχθούν Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την παρουσίαση. Κρίμα που δεν συμπεριλάβατε και το Πανεπιστήμιο του Σόνση, γιατί και εμείς έχουμε ένα δεύτερο κάμπους ε, και μάλιστα πρόκειται για ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και είμαστε ιδιαίτερη περήφανοι γι' αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω για την κατάσταση και τη σχέση με τις ε, τοπικές αρχές. Πρόσφατα το Κάρντιφ, που είναι η πρωτεύουσα της Ουαλίας, ε, ανακοίνωσε τεράστιες περικοπές στον προϋπολογισμό του πολιτισμού. Κάτι που θα ε, τροχοπεδίσει πολλά πολιτιστικά προγράμματα στην πόλη. Ευτυχώς βέβαια ανατράπει αυτή η προσπάθεια Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας των τοπικών αρχών, ε, ίσως με κάποιες ομίλους από τους κλάδους της δημιουργίας ε, και της τέχνης, ώστε να προωθηθούν σχέδια και προγράμματα, ε, ώστε να αποτραπούν τέτοιες καταστάσεις ή έστω και βραχυπρόθεσμα, να μην χρειαστούν να μην χρειαστεί να σταματήσουν προγράμματα ή να κλείνουν κινηματογράφοι εξαιτίας ε, των περικοπών που γίνεται στους κρατικούς προϋπολογισμούς ιδιαίτερα για θέματα πολιτισμού. Ε, κύριε Λιμπάτσκα, ευχαριστώ. Εγώ παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, περιμένω, περιμένω βάλετε τα ακουστικά σας, παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσίασή σας, γιατί σε μεγάλο βαθμό απάντηση στι ερωτήσει ε, που ε, υπέβαλα χθε στον Επίτροπο Ναύρατσιτς. Ρώτησα λοιπόν χθε ε, τον Επίτροπο με ποιον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνέργεια μεταξύ των, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του επενδυτικού σχεδίου του Juncker, τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς. Σε κάποιο βαθμό απάντησε χθε ο Επίτροπος και απαντήσατε και σήμερα και εσείς με την παρουσίασή σας. Έχω όμως κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις. Πώς μπορούμε να διευρύνουμε αυτή τη συνέργεια και να συνδυάσουμε τη συνεργασία και με τα διαστρωτικά ταμεία, με το Ταμείο Συνοχής και με προγράμματα όπως το ορίζοντας 2020. Γιατί αυτό που ε, δημιουργεί πρόσκομα στην Πολωνία τουλάχιστον για την ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο φόβος του κόστους του κινδύνου αυτού, του ρίσκου. Πώς θα γίνει ο καταμερισμός του κόστους, ε, του ρίσκου της αποτυχίας για παράδειγμα. Δεν μπορεί ο ειδικό κλάδος να αναλάβει μόνο αυτό το ρίσκο της αποτυχίας. Βλέπετε κάποια δυνατότητα να ενισχυθεί, ε, να ενισχυθούν τα αποτελέσματα σημαντικών ερευνητικών προγραμμάτων όπως το Ρίζοντας 2020 ή το Έρασμος, για παράδειγμα. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις διευθύνσεις που εκπροσωπούνται εδώ θα ήθελε το λόγο. Παρακαλώ. Thank you. Uh, I will start. I may have colleagues who... Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω εγώ και ίσως οι συνάδελφοι συμπληρώσουν στη συνέχεια αυτά που θα πω. Ευχαριστούμε κύριε Γκρουμπέρ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση που μας κάνατε maybe repeat a bit what, what... Και θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπατε, γιατί είδαμε τις ίδιες τάσεις στις συζητήσεις που είχαμε με τα κράτη-μέλη ε, και τους ε, κάποιων προγραμμάτων. Είχαμε το προηγούμενο Οκτώβριο μία ε, διάσκεψη με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με στόχο να ενημερώσουμε καλύτερα για τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που δίνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και να κινητοποιήσουμε ενδιαφερόμενους ώστε να ε, υποβάλουν προγράμματα και σχέδια. Και καταλήξαμε σε δύο συμπεράσματα από τη διάσκεψη αυτή. Ε, σε ό,τι αφορά την παιδεία, έχουμε πρόβλημα με τα πολύ μικρή εμβέλεια προγράμματα. Ε, υπάρχει εκεί πρόσκομα στη δημιουργία των προγραμμάτων. Αυτά τα μικρή εμβέλεια προγράμματα θα καταφέρουν να συνδυαστούν αυτό είναι πρόβλημα. Δεύτερο πρόβλημα είναι ε, το μείγμα κρατικής και ιδιωτικής ε, χρηματοδότησης. Μερικές φορές υπάρχουν και νομικά προσκόμματα για το συνδυασμό κρατικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης σε ορισμένες χώρες τουλάχιστον. Επίσης, ε, καταλήξαμε και σε ένα άλλο συμπέρασμα. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν ιδιωτικοποιεί την κρατική στήριξη της παιδείας. Όχι, απλώς τη συμπληρώνει, γιατί έχουμε χάσμα στις, στις υποδομές, κυρίως στην παιδεία και αλλού. Γι' αυτό θα πρέπει να κινητοποιήσουμε όσους πόρους έχουμε για να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα. Είναι συμπληρωματικό να τονίσουμε αυτή τη συμπληρωματικότητα μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών κονδυλίων. Πώς λοιπόν θα υπερκεράσουμε όλα αυτά τα εμπόδια. Αυτό που επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να εξετάσει διάφορες εναλλακτικέ λύσεις. Μία που θέλουμε να την αναλύσουμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι να συνδυάσουμε μικρά προγράμματα μέσω επενδυτικών πλατφορμών. Ακόμη δεν βρήκαμε τη λύση, αλλά το διερευνούμε για να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε να συνδεθούν όλα αυτά τα μικροπρογράμματα. Βέβαια θα πρέπει ε, να δραστηριοποιηθούν οι συντάκτες των σχεδίων και προγραμμάτων στην Αθηνά και χείρα εκείνη. Επίσης, ε, πολύ σημαντικό είναι αυτό το κέντρο, συμβουλευτικό κέντρο επενδύσεων, αυτό το advisory hub που είπατε για να γίνει καλύτερη προετοιμασία και βοήθεια της προετοιμασίας σε τοπικό επίπεδο. Και σε ό,τι αφορά τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα, Πολύ σημαντικό το σχόλιο σας, γιατί το Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει το θεματολόγιο για τις δεξιότητες, για να δούμε πώς θα συνδυάσουμε τα διάφορα μέτρα στήριξης ε, χρηματοδοτικά που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά το ΕΦΣΙ και το επιδετικό ε, πρόγραμμα, αλλά συνδυασμό τους και με τα διαρθρωτικά ταμεία, με το Ορίζοντα 2000, με το έρασμο ε, συν Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν το έργο που έχουμε μπροστά μας και φυσικά θέλουμε ευρεία εταιρική σχέση και συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να το υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Σύντομα παρακαλώ γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα από τη δική μας πλευρά, τη δική μας Γενική Διεύθυνση να ευχαριστήσουμε και πάλι τον κύριο Γκρούμπερ. Στις 10 Μαρτίου διοργανώνουμε εργαστήριο των stakeholder με συγκεκριμένους stakeholders. Θα έχουμε και εταιρείε και ενώσεις από τον ε, κλάδο των πνευματικών δημιουργών. Θα έχουμε και άλλους που ενδιαφέρονται και βεβαίως και συναδέλφους από άλλες γενικές διευθύνσεις, τη GD Connect για την ε, Guarantee Facility. Ε, θα είναι λοιπόν ένα εργαστήρι που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τα πράγματα αυτά. Έχουμε αρχίσει ήδη να συνεργαζόμαστε με ορισμένε ενώσει για μια ενδεχόμενη δημιουργία δέσμης διαφόρων πρωτοβουλειών. Είναι ιδέες που θα θέλαμε να δοκιμάσουμε και στην πράξη. Ήθελα να σας δώσω τις προφορίες αυτές για το σεμινάριο, για το εργαστήριο. Εγώ είμαι από την DG Connect να σας πω πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την Guarantee Facility του EIF. Βρισκόμαστε πια στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων και είμαστε πεπισμένες ότι θα μπορέσουμε να υπογράψουμε τη Συμφωνία Ανάθεσης πολύ σύντομα. Αρχίζουμε και επικοινωνιακές δράσεις προς τον τομέα μαζί με τις συναρμόδιες διευθύνσεις και κινητοποιούμε το Creative Europe Desk και όλα τα desk αυτά, όλα τα γραφεία αυτά <clears throat> τα οποία βρίσκονται σε διάφορες χώρες μέλη. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο όλο τον πολιτιστικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω να τονίσω το εξής. <clears throat> Δείξατε με ξεκάθαρο τρόπο ποια είναι τα εμπόδια, οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες. Είμαι σίγουρη μετά από τις παρεμβάσεις των συναδέλφων ότι χωρίς τον προδραστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την δημιουργία αυτής της πλατφόρμας δεν θα βοηθηθούν οι επιχειρήσεις με επαρκή τρόπο. Θέλουμε λοιπόν οι προτεραιότητες αυτές να μην αγνοηθούν από άλλους τομείς που πολλές φορές οι άλλοι τομείς έχουν το βάρος να επιβάλλουν και να στρέψουν τις απόψεις τους και να στρέψουν την προσοχή των επενδυτών προς αυτές. Δύο ερωτήσεις εδώ λοιπόν. Δημιουργείται ένα πόρταλ στο διαδίκτυο είπατε στο οποίο θα μπαίνει κανείς εύκολα για να δούμε ποια είναι τα προγράμματα τα οποία είναι διαθέσιμα και ένα πόρταλ το οποίο θα πρέπει να είναι και πληροφοριακό. Δηλαδή, πέρα από τις διαδικασίες ευαισθητοποίησης, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Και δεύτερη ερώτηση, οι επενδύσεις οι οποίες έρχονται είναι ευρωπαϊκές επενδύσεις ή ζητάτε και από οικονομικούς εταίρους εκτός Ένωσης να δραστηριοποιηθούν. Έχω την αίσθηση ότι το θέμα αυτό δεν τελειώνει ε, βέβαια εδώ. Νομίζω ότι η αρχική πρόταση είναι πολλά υποσχόμενη. Vanno tenuti presenti perché sono promettenti in termini eh, diciamo, di crescita, di occupabilità e anche naturalmente di coesione sociale, quindi questi hanno un Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναζητήσουμε για να βελτιώσουμε ε, την προστιθέμενη αξία ε, της ε, παρέμβασης της επενδυτικής. Είναι σημαντικό πάντως το ότι σήμερα είναι υπομελέτη το νέο χρηματοδοτικό μέσο Αναφέρομαι όμως κυρίως σε θέματα πνευματικής ε, δημιουργίας. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο το ΕΦΣΙ, το στρατηγικό πρόγραμμα, θα ανοίξει νέες προοπτικές. Ε, έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μας. Σας δίνουμε το λόγο λοιπόν για να μας παρουσιάσετε τα συμπεράσματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Ε, θα παρουσιάσω τις απαντήσεις μου με τη σειρά που τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο για την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού έργου. Χρειάζεται να γίνει διάκριση ποιο είναι το πρόγραμμα διδασκαλίας και ποιο άλλο το ένα λοιπόν και άλλο η υποδομή και βλέπουμε κυρίως στον ιδιωτικό τομέα να κάνει επενδύσεις στις υποδομές, κτηριακές υποδομές και άλλες. Εκεί έχει και ε, το πλεονέκτημα ο ιδιωτικό τομέας. Αυτό ίσως να αλλάξει βέβαια κάπως ίσως στον τομέα της ε, ανώτατης εκπαίδευσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, οπότε ίσως είναι χρήσιμο να υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στο περιεχόμενο αν αλλάξω μικρόφωνο, ε, εκεί όπου ο ιδιωτικός τομέας έχει ε, καλή ε, γνώση είναι στην επαγγελματική κατάρτιση. Αλλά έχουμε υπόψη μας τις ανησυχίες αυτές. Το πρόγραμμα ΕΦΣΙ τώρα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, κατά πόσο ασχολείται με τις λεγόμενες δημιουργικές δημιουργικούς τομείς, τομείς της πνευματικής δημιουργίας. Υπάρχει εκεί πραγματικά ευρύ πεδίο ε, να ε, δοθούν δάνεια και σε αυτό τον τομέα. Όμως επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για το εάν ε, θα είναι δυνατόν και εκεί αυτό το, ο συμβουλευτικός άξονας το advisory hub θα είναι χρήσιμο νομίζω. Υπάρχει ακόμα πολύ ανάγκη για υποδομές. Η τράπεζά μας έχει μεγάλη εμπειρία στην χρηματοδότηση υποδομών, για παράδειγμα αιθουσών ε, συναυλιών ε, που καμιά φορά εντάσσονται και στα πλαίσια της ε, ανακαίνησης αστικών κέντρων και συχνά για παράδειγμα φανταστείτε την ανακαίνιση μιας όπερας τι συμβαίνει όλο αυτό για τους διάφορους τομείς και κλάδους που είναι συναρμόδιοι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σας το έδειξα και στον πίνακα, είναι η βασική συνεισφορή στην επίλυση του προβλήματος της εκπαιδεύσεως. Η Ευρώπη έχει έναν πολύ ισχυρό τομέα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρξουν οι σωστές δεξιότητες έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να απορροφούν τους νέους που ζητούν δουλειά είναι ξεκάθαρο ότι ο βασικό συνεισφορέα για τη λύση του προβλήματο είναι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Για το Σόνσι είναι καλό το παράδειγμά σα. Είχαμε μάλιστα και case study όταν κάναμε το σεμινάριό μας, σεμινάριό μας όπως είπε και η κυρία Έριξον. Είναι καλό παράδειγμα αυτό που αναφέρατε και καλό παράδειγμα μιας μετατροπής ενός ε, βιομηχανικού τοπίου σε ε, βιομηχανικού χώρου δηλαδή, ε, σε ε, πανεπιστημιακές σχολές. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά που θα έδειχναν ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του Εύση στον τομέα της εκπαιδεύσεως. Υπάρχουν πολλές ανάγκες σχετικά. Εγώ έχω δει πολλές χώρες έχουν να δείξουν όπως το Λουξεμβούργο για παράδειγμα που πήρε κτίρια της Χαλιβουργίας και τα έχει μετατρέψει σε πανεπιστημιακές σχολές. Στην Ιταλία το ίδιο. Έχουν πάρει ε, ε, παλαιότερες δραστηριότητες και τις έχουν μετατρέψει σε δραστηριότητες που εξυπηρετούν τον ε, σύγχρονο αιώνα. Τώρα, το αποτέλεσμα συνεργειών υπάρχει ακόμα πεδίο. Το εύση το ίδιο είναι ακριβώς ένα παράδειγμα των συνεργειών που μπορεί να επιτύχει κανείς. Και μέσα στο ΕΦΣΥ υπάρχει περιθώριο και το αναπτύσσουμε, δηλαδή για παράδειγμα προσπαθούμε να φτιάξουμε equity funds που θα έχουν ως στόχο να χρησιμοποιήσουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον χώρο για παράδειγμα των διαφθορτικών ταμείων. Έχετε συχνά το πρόβλημα επειδή δεν είναι ένας φορέας τράπεζα προχωρείται στην δημιουργία του έργου αλλά χρειάζεται και παρακολουθή του. Άρα ενδέχεται κάποιο επίπεδο χρέωσης να είναι χρήσιμο για την μακροπρόθεσμη δημοσιονομική πειθαρχία του έργου. Αυτά. Αυτά νομίζω έληξε ο χρόνος μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρο ε, Σίλβα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σα, για την ευκρίνεια γενικά των λεγόμενων σας. Είναι μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Επιτροπή αλλά και την τραπεζά σας. Υπολογίζουμε λοιπόν στην δική σας παρουσία και προσωπικά ε, ε, τη δική σας ε, συμμετοχή κύριε Γκρούμπερ να αυξήσουμε την ευαισθησία η οποία απαιτείται ε, για τον τομέα έτσι ώστε να ευνοήσουμε ακριβώς αυτό τον συνδυασμό των διαφορετικών εμπειριών μας. Η εκστρατεία αυτή η πληροφόρηση θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ε, βάρος και για τη δική μου χώρα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, ευχαριστώ και την Επιτροπή και τους συναδέλφους. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον αγαπητοί συνάδελφοι, δηλαδή την παρουσίαση μιας μελέτης σε μια στρατηγική στιγμή θα έλεγα. Καλώς ήρθατε. take your για το θέμα λοιπόν των Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Πολιτισμού στο εξωτερικό. If you can, uh, sorry. A little silence, please. Sorry, because we have to continue our work. Λοιπόν, πρέπει να συνεχίσουμε λίγη ησυχία, παρακαλώ. Ευχαριστώ λοιπόν τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσία τους. Καλωσορίζω και τις ε, ερευνήτριες, την κυρία Σμιτ και την κυρία Ντεμπεφ. Οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν την έκθεσή του. στόχο της συγκεκριμένης μελέτης είναι να υπάρξει καλύτερη κατανόηση του στρατηγικού ρόλου και του συντονισμού του ρόλου αυτού ε, από πλευράς της Ένωση και των κρατών μελών σχετικά με την προώθηση του πολιτισμού προς τρίτες χώρες. Είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι έχει ανακοινωθεί μια νέα στρατηγική για τη λεγόμενη ε, πολιτιστική διπλωματία. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια κάποια μορφή διαλόγου για τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Η Επίτροπος μας είπε ότι θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία τον επόμενο μήνα μαζί με τον Επίτροπο για τη Διεθνή Συνεργασία και την ε, ε, είπατε εκπρόσωπο. Λοιπόν, πρέπει να μας πείτε σήμερα, να μας δείξετε σήμερα ποιες είναι οι σωστές πρακτικές και οι σωστές εμπειρίες και τα μοντέλα συνεργασίας και συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον να τα ακούσουμε. Και ήδη τα Εθνικά Ινστιτούτα Πολιτισμού είναι ένας εταίρος που με τη σειρά του θα μπορούσε να βοηθήσει στον συνδυασμό των εμπειριών που υπάρχουν για την προώθηση της πολιτιστικής ταυτότητας και για τους διαπολιτιστικούς δεσμούς με τις τρίτες χώρες. Έχουμε, πρέπει να κλείσουμε αυτό το κομμάτι πριν τις 11. Έχουμε λοιπόν κάποιο χρόνο να προχωρήσουμε. Έχετε το λόγο κυρία Σμιτ, κυρία Ντομπέφ. Σας ευχαριστώ κυρία Κώστα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη γραμματεία της Επιτροπής για την ευκαιρία που μας έδωσε να καταρτήσουμε, να εκπονήσουμε αυτή τη μελέτη και να σας την παρουσιάσουμε σήμερα. Όπως είπε και η πρόεδρος ε, Κώστα, είναι πολύ επίκαιρη αυτή η μελέτη γιατί εκπονήθηκε τη στιγμή που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονήθηκε τη στρατηγική για την ε, πολιτιστική διπλωματία, τη διπλωματία μέσα των πολιτιστικών σχέσεων όπως αναφέρεται. Η κυρία Μογκερίνη μάλιστα θα υποβάλει και νέα ανακοίνωση ε, στο ε, επικείμενο πολιτιστικό φόρουμ που θα λάβει χώρα φέτος τον Απρίλιο. Η μελέτη μας ε, δημοσιεύθηκε πριν από δύο εβδομάδες στον ιστότοπο της Επιτροπής σας και έκτοτε λάβαμε πολύ θετικά σχόλια, ιδιαίτερα από τους πολιτιστικούς οργανισμούς πολλά τέτοια πολιτιστικά αισθητήτα και οργανισμοί μας επισήμαναν ότι η μελέτη είναι πολύ σημαντικό βήμα στην προσπάθεια δημιουργίας νέου επίπεδου ευρωπαϊκών πολιτιστικών σχέσεων. Ήταν πολύ χρήσιμη η μεγάλη απήχηση που είχε η μελέτη και το ζωηρό ενδιαφέρον που δημιούργησε. Να σας παρουσιάσω συντομία τη μελέτη μας. Αναλύει καταρχήν το ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι πολιτιστικοί οργανισμοί στην ευρωπαϊκή στρατηγική ή την πολιτιστική. Αναλύσαμε τις ε, δομές αυτών των ε, οργανισμών και αισθητούτων και κατά πόσο οι δραστηριότητες τους έχουν ήδη μια ευρωπαϊκή διάσταση ή κατά πόσο θα μπορούσε να ενισχυθεί ή να αξιολογηθεί ο ρόλος που θα μπορούσαν να παίξουν. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε τους 29 πολιτιστικούς οργανισμούς που εξετάσαμε από 22 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μερικές περιπτώσεις ε, έχουμε περισσότερα από ένα από πολιτιστικούς οργανισμούς στα κράτη-μέλη για πολιτικούς ιστορικούς λόγους υπάρχει περισσότερο από ένα τέτοιο Ινστιτούτο η ιδέα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τον πολιτισμό και τις εξωτερικές σχέσεις δεν είναι καινούρια. Ε, και μάλιστα εκπορέθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή η ιδέα της στρατηγικής ε, της, ε, της πολιτιστικής διπλωματίας. Αν δεν κάνω λάθος, το 2011 ψηφίστηκε ένα ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τέτοια πρόταση και αποτέλεσε τον εναρκτήριο λακτίσμα κάποιων προκαταρκτικών δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διενεργήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με ένα όμιλο πολιτιστικών οργανισμών και μια εταιρεία συμβούλων. Αυτές οι προκατακτικές δράσεις για την πολιτιστική διπλωματία είναι πολύ σημαντικές γιατί δείχνουν ότι και οι τρίτες χώρες είναι έτοιμες να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον πολιτιστικό τομέα. και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ο σύνολο και με τα επιμέρους κράτη-μέλη θέλουν συνεργασία οι τρίτες χώρες. Πολύ ενθαρρυντικό. Ε, μάλιστα η μελέτη μας περιλαμβάνει και κάποιες ε, πρακτικές στάσεις για το πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε οι προκαταρκτικές αυτές ε, δράσεις αποτέλεσαν έμπνευση για πολλές άλλες δραστηριότητες που ε, λήφθησαν από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και από το Κοινοβούλιο. Και μάλιστα στην Επιτροπή Πολιτισμού συζητήθηκε σε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αυτό το θέμα. Και μάλιστα και στη γνωμοδότηση της κυρίας Γουόρντ αναφέρθηκε η προπαρασκευαστική αυτή δράση που ξεκίνησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως σας είπα. Τώρα, τι συνέχεια δόθηκε σε αυτή την προκατακτική δράση. Νομίζω ότι αυτός ο τρόπος σκέψης είναι σημαντικός. Ε, να χρησιμοποιήσουμε τα πολιτισμικά μας ε, ατού στη διπλωματία. Έτσι ενισχύουμε το πολιτικό μας βάρος και βελτιώνουμε τις σχέσεις μας με τις άλλες χώρες. Σχέσεις που στηρίζονται σε αμοιβαία κατανόηση, σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και δημιουργούν καλύτερη εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό. Και όταν μιλούμε για τον πολιτισμό, για τις πολιτιστικές σχέσεις και την πολιτιστική διπλωματία, εκλαμβάνουμε τον πολιτισμό με την ευρία έννοια, διασταλτικά. Καλύπτουμε τον τομέα της δημιουργίας, τον αθλητισμό, την παιδεία, την κοινωνία των πολιτών, αλλά και ε, τις κοινέ αξίες, τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά είναι τμήμα της κουλτούρας μας. Και όταν μιλούμε για ευρωπαϊκή πολιτιστική διπλωματία, προσπαθούμε να βρούμε νέους τρόπους συσχετισμού με τις ε, τρίτες χώρες. Ε, θέλουμε να ενισχύσουμε τις διαπροσωπικές επαφές, ε, την πρόθεση κοινών προγραμμάτων και σχεδίων, την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και του διαλόγου. Και αυτό δεν γίνεται μόνο με εκδηλώσει όπου το κάθε Ινστιτούτο, κάθε πολιτιστικό οργανισμό προωθεί τη δική του κουλτούρα και το δικό του πολιτισμό, αλλά ε, δίνεται μια ευρωπαϊκή διάσταση και μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θα δώσω τώρα το λόγο στη συνάδελφο τη Κλιμεντίν, που θα μα μιλήσει για τι διάφορε δομέ τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και θα τονίσει την ευρωπαϊκή ε, διάσταση αυτών των δραστηριοτήτων. Σα ευχαριστώ, Γιολάντα εξετάζουμε τις ιδιαιτερότητες των ε, πολιτιστικών Ινστιτούτων υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεταξύ τους και σε ό,τι αφορά το μέγεθος και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διοίκησή τους, την προώθηση των ε, ε, ευρωπαϊκών ιδεών και τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά project. Παρά τις διαφορές έχουν παρόμοια αποστολή, δηλαδή την προώθηση του πολιτισμού και να δείξουν την ε, ε, ζωτικότητα της καλλιτεχνικής κοινής στις διάφορες χώρες. Σε ό,τι αφορά το τι πράττουν στο εξωτερικό βλέπουμε ότι έχουν ε, κοινά δίκτυα με αξία 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό το έργο παράγεται κυρίως από τα μεγάλα βέβαια ιδρύματα, είναι παρόντα σε 156 χώρες εκτός της Ένωσης, έχουν 30.000 ε, προσωπικό και 2.170 γραφεία. Ε, ξεφεύγουν από την ε, άμεση σφαίρα επιρροής των χωρών τους και βάζουν περισσότερο στρατηγικές κατευθύνσεις την ανατολική και στην νότια γειτονία αυτή η δραστηριοποιείται κυρίω και αυτό απηχεί και τις νέες θεματικές τους προτεραιότητες αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης των νέων μεταναστευτικό, προσφυγικό διαπολιτιστικός και διαθρησκιακός διάλογος ε, ακολουθώντας και τις ε, σύγχρονες προτεραιότητες Τώρα η ευρωπαϊκή διάσταση αυτών των πολιτιστικών ιδρυμάτων δεν έχουν αρητή εντολή ούτε στην ε, αποστολή τους να προωθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ε, θεμελιώδεις αξίες της, ωστόσο μέσα από συγκεκριμένες δράσεις το πράττουν. Τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα ε, συμμετέχουν σε δύο μεγάλα δίκτυα, το UNIC, το οποίο ανέφερε προηγουμένως ο συναδελφός μου, που είναι ένα σχετικά νέο, μόλις δεκαετών δίκτυο και έχει ε, το βασικό του γραφείο στις Βρυξέλλες. Το Γιονίκ είναι νεαρός φορέας. Ήδη προωθεί μια στρατηγική για να οργανωθεί καλύτερα και να παίξει κέριο, κέριο ρόλο σε αυτή την ε, στρατηγική για την πρόθεση των, ε, των ευρωπαϊκών ειδών. Και ε, το άλλο είναι το προ το οποίο να έχει παρόμοιους στόχους. Ορισμένα πολιτιστικά ιδρύματα έχουν γραφεία στις Βρυξέλλες, τα οποία ήταν σε επαφή μαζί μας, αλλά διατηρούν και επαφές με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να γνωρίζουν τι συμβαίνει, αλλά και για να έχουν και πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και έχουμε και τα κλάστερα αυτά, τα κέντρα, είναι 95 συνολικά, 50 σε τρίτες χώρες, δεν είναι πλήρως οργανωμένα και λειτουργικά όλα αυτά τα κλάστερ, αλλά μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για να προσθέσουν την ευρωπαϊκή διάσταση στις πολιτιστικές τους δραστηριότητες. Αυτά τα κλάστερ του UNIC με φέρνουν στο επόμενο θέμα μου, που είναι δηλαδή έργα, project, ε, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο δίκτυο το οποίο έχει τη σχετική ικανότητα αλλά και τεχνογνωσία για να ηγηθεί σε αυτά τα έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Παίζουν ένα στρατηγικό ρόλο. Εδώ έχουμε δύο ενδιαφέροντα παραδείγματα κλάστερ του UNIC που συνεργάζονται με τη, σε, χέρι με χέρι με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία στην Ιορδανία και στην Τινησία. Και στην Τινησία μάλιστα το κλάστερ αυτό, το κέντρο αυτό έχει λάβει ένα σημαντικό προϋπολογισμό για να προωθήσει ένα πολιτιστικό πρόγραμμα μαζί με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία εκεί για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού της Ισίας. Να επιστρέψω το μικρόφωνο στη συνάδελφό μου που θα εξηγήσει ποια είναι τα ισχυρά σημεία και ποια είναι τα αδύναμα σημεία. Πώς μπορούν τα πολιτιστικά ιδρύματα να εξυπηρετήσουν τη νέα πολιτική για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, εξετάσαμε τα ισχυρά και τα λιγότερα ισχυρά σημεία τους, τις ευκαιρίες που δημιουργούν και προσφέρουν, αλλά και τις απειλές, υπάρχουν και απειλές που τα απειλούν. Έχουμε δει ότι τα πολιτιστικά ιδρύματα προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αντισταθμίσουν τις αδυναμίες των ευρωπαϊκών θεσμών. Ε, για παράδειγμα, την έλλειψη πλήρους αρμοδιότητας ε, για απασχόληση με πολιτιστικά θέματα, αλλά και δεν έχουν και επαρκή πείρα οι ευρωπαϊκές Αντιπροσωπείς ανά τον κόσμο για να ασκήσουν την πολιτιστική διπλωματία. Ε, υπάρχουν περίπου 140 αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο και πολύ λίγες, νομίζω μόνο τρεις έχουν εκεί και κάποιον ο οποίος ασχολείται με τον ε, πολιτισμό. Οι υπόλοιπε δεν έχουν κάποιον ειδικό για τα πολιτιστικά θέματα. Συνήθω τα αναλαμβάνει ο αρμόδιος για ε, επαφέ με τον τύπο ή τα μέσα γενικώ. ή σε συνεργασία με τα πολιτιστικά ιδρύματα. Ποια είναι τα ισχυρά τώρα σημεία των πολιτιστικών ιδρυμάτων. Μία από αυτές, ε, μία από αυτά, ένα από αυτά τα ισχυρά σημεία είναι ότι διαθέτουν τους πόρους. Ε, ε, προσφέρουν τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκμεταλλευτεί τα ισχυρά αυτά σημεία, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη να δημιουργήσει επικαλυπτόμενες εν τέλει δομές. Και τα δίκτυα βεβαίως. Επειδή πολλά από αυτά τα πολιτιστικά ιδρύματα υπάρχουν και λειτουργούν εδώ και πολύ καιρό, ορισμένα μάλιστα ήδη έχουν κλείσει την 70η ετία, πριν ακόμα να υπογραφεί η Έχουν λοιπόν την ευκαιρία, ή είχαν την ευκαιρία, να δημιουργήσουν παγκόσμια δίκτυα με συνεργασία φορέων της κοινωνίας των πολιτών σε τρίτες χώρες, με συνεργασία των κυβερνήσεων, για να ασχοληθούν με θέματα πολιτιστικά και άλλα σχετικά και βέβαια και με τους πολιτιστικούς φορείς στις ε, ε, χώρες όπου δραστηριοποιούνται και βεβαίως έχουν και καλή διασύνδεση με τις ευρωπαϊκές αντιπροσωπείες, τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα ιδρύματα αυτά θεωρούνται αξιόπιστοι εταίροι για τον κόσμο στις τρίτες χώρες και δεν έχουν έτσι, δεν δίνουν την εικόνα προπαγανδιστικών μηχανισμών της κυβέρνησης. Αυτό είναι σημαντικό. Σήμερα ιδίως όπου αντιμετωπίζουμε πολλές δυσκολίες λόγω των ε, κρίσεων ανά τον κόσμο και όπου ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας δεν είναι απαραίτητα ο καλύτερος. Χρειάζεται λοιπόν να ψάξουμε να βρούμε καινούριου τρόπους για να, ε, να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο και τις κοινωνίες εκεί τοπικά. Το άλλο είναι η τεχνογνωσία. η επικεφαλής των αντιπροσωπιών έχουν γνώση και στρατηγική τεχνογνωσία και μπορούν να προσφέρουν συμβουλές στους ευρωπαϊκούς θεσμούς σχετικά με τη στρατηγική που θα πρέπει να εφαρμόζουν. Διαθέτουν τεχνογνωσία δηλαδή και στην ανάπτυξη πολιτιστικών έργων αλλά και ορισμένων ευρωπαϊκών. Τώρα ποια είναι τα αδύναμα σημεία των πολιτιστικών ιδρυμάτων. Εδώ τονίζω ένα βασικά δεν έχουν εντολή. Δεν διαθέτουν εντολή. Τα περισσότερα πολιτιστικά ιδρύματα έχουν ειδική εντολή να προωθούν τον εθνικό πολιτισμό των χωρών από τις οποίες προέρχονται. Με κάποιες εξαιρέσεις, στο λεγόμενο mission statement δεν αναφέρονται σε ευρωπαϊκές δραστηριότητες ή δραστηριότητες σχετιζόμενες με την Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει διότι αν δεν περιλαμβάνεται στο mission statement πάει να πει ότι δεν μπαίνει και στο πρόγραμμα εργασιών τους. Αν δεν μπαίνει στο πρόγραμμα εργασιών τους δεν ε, διατίθενται πόροι αλλά ούτε και προσωπικό. Γι' αυτό φτάνει πια το ευρωπαϊκό γίγνεσθε σχόλιο να μπαίνει τελευταίο στις προτεραιότητες τους. Ποιε είναι οι ευκαιρίες τώρα. Μια από τις μεγάλες ευκαιρίες που διαπιστώσαμε εμείς είναι ότι πολλά από τα πολιτιστικά ιδρύματα έχουν την διάθεση να ευθυγραμμίσουν τις ε, γεωγραφικές και θεματικές τους προτεραιότητες με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμούς στρατηγικούς εταίρους και στις γειτονικές της χώρες. Και τα πολιτιστικά ιδρύματα ε, στηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Απειλές. Υπάρχει ένας αριθμός απειλών Μία που επιθυμώ να τονίσω ιδιαίτερος είναι η μονοπόληση από τα μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα τα οποία είναι 4 έως 7 όπως θέλετε έχουν μεγάλους προϋπολογισμούς, πολλά γραφεία και αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μονοπολίσουν τον προϋπολογισμό που είναι διαθέσιμος για τέτοιες εξωτερικές δραστηριότητες. Άρα μειώνονται οι ευκαιρίες για άλλους πολιτιστικούς φορείς οι οποίοι έχουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν. Συστάσεις. Ναι, θεωρούμε ότι μπορούν να παίξουν ένα ρόλο τα ιδρύματα αυτά, διότι ήδη εκτελούν έργα και νομίζουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολο της και οι χώρες μέλη μπορούν να υποφεληθούν εάν ε, συμβάλλουν στη δημιουργία δεξαμενών τεχνογνωσίας και προσωπικού. ώστε να προσφέρουν και μεγαλύτερη ορατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο έργο που κάνει σε τρίτες χώρες. Για να δημιουργηθεί η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των πολιτιστικών διδρυμάτων, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διέπονται από ορισμένε αρχές. Η πρώτη θα πρέπει να είναι να, ζητηθούν, να ζητηθεί από τις κυβερνήσεις να χορηγήσουν εντολή στο πολιτιστικό ίδρυμα να ασχοληθεί με ευρωπαϊκά θέματα. Άρα, ρητή εντολή, για να είναι σαφές. Δεύτερο, όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να εκτελούνται μέσα στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής δράσης που ανέφερα προηγουμένως δηλαδή προώθηση ε, προγραμμάτων στην βάση της συνεργασίας. Τρίτο, πολύ σημαντικό νομίζω, ως σύσταση εννοώ, είναι για να γίνονται σεβαστές ορισμένες υποχρεώσεις τα πολιτιστικά ιδρύματα στα οποία θα ανατεθεί μια ευρωπαϊκή αποστολή θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να υπογράψουν ένα μνημόνιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων που θα προβλέπει ξεκάθαρα ποιε είναι οι υποχρεώσει των συμβαλωμένων μερών. Τέταρτη σύσταση, την οποία τονίζω ιδιαίτερα, τα πολιτιστικά ιδρύματα θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συνεργαστούν με άλλε μη κρατικές οργανώσει και με δημόσιου φορεί, ούτω ώστε να ενθαρρυνθεί η εμπλοκή ή πάντως να δημιουργηθούν πανευρωπαϊκά δίκτυα και να εξασφαλιστεί ότι και άλλοι φορείς θα μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δημιουργώντας έτσι ένα πολλαπλασιστικό αποτέλεσμα. Να δοθούν και κίνητρα στα πολιτιστικά ιδρύματα μέσω διαβούλευσης, ε, με χρηματοδοτική στήριξη. διάρκεια που έχουν ευρωπαϊκή διάσταση, που σημαίνουν προώθηση ευρωπαϊκών αξιών και για να δημιουργηθεί και μεγαλύτερη διαφάνεια και έτσι ώστε οι διαδικασίες να είναι ανοιχτές και διαφανείς, θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τρία κριτήρια επιλεξιμότητας εφόσον τα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το πολιτιστικό ίδρυμα θα πρέπει να δείχνει ότι έχει την ικανότητα να συνεργαστεί. Δεύτερο, να διασφαλίζεται ότι υπάρχει ισορροπία μεταξύ μικρών, μεγάλων και μεσαίων πολιτιστικών ιδρυμάτων γιατί θα πρέπει να εμπλέκονται και τα μικρά, όχι μόνο τα μεγάλα και τέλος να μπει και μία ρήτρα που να λέει ότι όσο αυτό είναι δυνατόν θα πρέπει να αναθέτουν υπεργολαβικά τις δραστηριότητες επιτόπου. Τελευταίο, τελευταίο θέμα, γιατί η πρόεδρος μου δίνει μόνο δύο λεπτά ακόμη έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει τη νέα στρατηγική έχουμε ε, στοχεύσει και σε ορισμένα πιλωτικά σχέδια για να δούμε τι μπορεί να αποδώσει και τι όχι είδαμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια στρατηγική που να είναι κατάλληλη για όλους θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις διάφορες περιφέρειες. Αυτό που συζητήσαμε με τα πολιτιστικά ιδρύματα μα έδειξε ότι ενδιαφέρονται πολύ να συνεργαστούν με τους ευρωπαϊκούς θεσμού σε χώρες όπου υπάρχουν δυσκολίες και όπου είναι περίπλοκα τα πράγματα. Τονίζω ένα πιλωτικό πρόγραμμα, η δημιουργία ενός οίκου τη Ευρώπης στο Ιράν. Γνωρίζετε το Ιράν ε, βρίσκεται σε φάση ανοίγματο και δείχνει διάθεση να συνεργαστεί και να αναπτύξει πολιτιστικές σχέσεις με άλλες χώρες. Για την ώρα μονάχα ένα πολιτιστικό ίδρυμα έχει γραφείο στην Τεχεράνη. Το Αυστριακό Πολιτιστικό Ίδρυμα. Δεν υπάρχει ούτε η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα να μια καλή ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός οίκος όπου θα συνέρχονται τα πολιτιστικά ιδρύματα και θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες τους ντόπιου να κάνουν ε, να αναλαμβάνουν δραστηριότητε σε συνεργασία με άλλους φορείς εκεί και ούτω καθεξής. Νομίζω να αρκεστώ σε αυτά κυρία Πρόεδρε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητή κυρία. Νομίζω έχουμε τις προϋποθέσεις τώρα για να εμβαθύνουμε το θέμα. Νομίζω ότι και το ότι αναλύσατε γύρω στα 30 Ινστιτούτα και πραγματικά είδατε και ποια είναι τα βασικά κεφάλαια των δραστηριοτήτων των Ινστιτούτων αυτών, τα θέματα της χρηματοδότησης από το δημόσιο, τα θέματα των σχέσεων μεταξύ τους και νομίζω ότι ήταν σαφές αυτό το οποίο μας είπατε και για τις αδυναμίες και τα ισχυρά του σημεία. Οι εμπειρίες οι οποίες υπάρχουν μέχρι τώρα τις γνωρίζουμε. Υπήρξε ένα πιλωτικό πρόγραμμα από πλευράς μας στο λεγόμενο More Europe στα πλαίσια του UNIC και νομίζω ότι ο ρόλος αυτός μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής διπλωματίας και με ενδιέφερε το γεγονός ότι στην παρούσα φάση τα Ινστιτούτα δεν έχουν στα πλαίσια της παρούσης εντολής τους κάτι το σαφές, ε, κάτι το οποίο πραγματικά να ε, μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση ε, των πολιτιστικών χαρακτηριστικών των χωρών τους. Είναι σημαντικό αυτό, όπως σημαντικές είναι και οι συστάσεις σας. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους που τον ζήτησαν αν τον ζήτησαν. Σβέρ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά τις καλεσμένες μας για την παρουσίασή τους. Έχω μία ερώτηση. Ποιες είναι οι θεμελιώδεις ε, οικουμενικές αξίες τις οποίες ε, θα πρέπει να στηρίζεται ο διαπολιτισμικός διάλογος γιατί δεν ήταν ε, οι αξίες που μας είπατε εσείς, οι πρωταρχικές ε, αξίες ε, του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Άλλος κανείς? Θα ήθελα να απαντήσετε αργότερα και ίσως να φωτίσετε κάποια άλλα σημεία της μελέτης και να μου πείτε τι δυνατότητα έχουν είτε μεμονωμένοι πολιτιστικοί οργανισμοί είτε δίκτυα τέτοιων πολιτιστικών Ινστιτούτων ε, για πρόσβαση σε κοινοτικά κονδύλια. ώστε να αποφύγουμε οι μεγάλοι εμβέλειες πολιτιστικοί οργανισμοί να μονοπολίσουν την κοινωτική χρηματοδότηση. Είπατε ότι ε, δεν, έχουν όλες, δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες πολιτιστικοί οργανισμοί. Ε, δεν θα πρέπει να ενισχύσουμε το συντηρησμό και να προωθήσουμε κοινέ δράσεις, γιατί μας μιλήσατε για το Ιράν και για άλλες χώρες και είπατε ότι ίσως σε αυτές τις χώρες ακόμη και δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι σημαντικοί πολιτιστικοί οργανισμοί να προωθήσουν τέτοιες πολιτιστικές δράσεις και σε αυτές τις χώρες ώστε να γίνουν οι πολιτιστικοί οργανισμοί μας σε τρίτες χώρες ένα είδος ε, Ευρωπαίων πρεσβευτών, πρεσβευτών της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Πιστεύετε ότι οι εθνικοί πολιτιστικοί οργανισμοί είναι έτοιμοι να κάνουν αυτό το ποιοτικό άλμα, να δώσουν μια πιο ευρωπαϊκή διάσταση στις πολιτιστικές τους δράσεις, να περιλάβουν και την ευρωπαϊκή διάσταση στις δράσεις τους. Πιστεύετε ότι είναι έτοιμοι οι οργανισμοί να κάνουν αυτό το βήμα. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Για τις ευρωπαϊκές αξίες. Όταν μίλησα για ευρωπαϊκές αξίες ε, αναφέρθηκα και εννοούσε τις αξίες που κατοχυρώνονται στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αξίες των άρθρων 3 και 21 συγκεκριμένα. Εκεί αναφέρονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η οικουμενικότητα και ο διέρετος χαρακτήρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αρχή της ισότητας, αλληλεγγύης, σεβασμός των αρχών του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Είναι σημαντικές και κατοχυρώνονται, παραλαμβάνω, στη συνθήκη αυτές τις αρχές εννοούσα όταν είπα για θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, Επανέρχομαι στο σχόλιο σας για τα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των πολιτιστικών οργανισμών. Το, συζητήσαμε αυτό το θέμα με τους πολιτιστικούς οργανισμούς και μας είπαν ότι προτιμούν να ε, ευέλικτα και πολυδιάστατα μοντέλα και πρότυπα συνεργασίας. Δεν θα πρέπει όλοι οι πολιτιστικοί οργανισμοί μιας χώρας να εμπλέκονται, αλλά εκείνοι που ενδιαφέρονται περισσότερο και φυσικά έχουν και τη δυνατότητα τέτοια συμμετοχή. Τέτοια πολυεπίπεδη και ευέλικτη συνεργασία προτιμούν. Στην περίπτωση της Τινησίας, για παράδειγμα, έχουμε πέντε ή έξι, αν δεν κάνω λάθος, πολιτιστικά Ινστιτούτα ε, που συμμετέχουν, τα μικρότερα όχι γιατί δεν έχουν γραφεία τους εκεί. Μέσω του σχεδίου αυτό όμως, μέσω αυτού του project, ε, εμπλέκονται και σε μια χώρα που κανονικά δεν έχουν, στην οποία δεν έχουν πολιτιστική προσφορά. Πρόκειται για ένα μεικτό μοντέλο. Δεν χρειάζεται όλοι να είναι παρόντες σε μια δεδομένη χώρα. Είναι παρόντες αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο και μέσω του project μπορούν να συμμετέχουν και οι μικρότεροι πολιτιστικοί οργανισμοί, εφόσον ε, παραλαμβάνουν ενδιαφέρονται. Και στο Ιράν συμμετέχουν εκείνοι που ενδιαφέρονται. Δεν υπάρχει υποχρέωση για όλους τους πολιτιστικούς οργανισμούς να δώσουν το παρόν. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι είχαμε διήμερη πολύ έντονη συνεδρίαση με υπερπλήρες πρόγραμμα και υπάρχει κάποια κόπωση. Αυτό δεν δείχνει όμως ε, έλλειψη ενδιαφέροντος, γιατί πραγματικά η μελέτη σας είναι πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Θέλετε να επανέλθετε κυρία Σβέρ, παρακαλώ. Έχω μια ερώτηση. Αναφέρονται μερικές αξίες ως ε, προσπάθεια προώθησης των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών αφαίνοντας τις διαφάνειες, αλλά στις διαφάνειες δεν, δεν περιλήφθησαν τα θεμελιώδη δικαιώματα που μας αναφέρατε προηγουμένως. Υπάρχει διαφορά λοιπόν. Φαντάζομαι όμως ότι θα τηρήσετε και θα τιμήσετε τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καταχαιρώνονται στις συνθήκες, εννοείται. Φυσικά, βεβαίως. Όταν μιλούμε για θεμελιώδεις αξίες, ε, δεν μπορούμε να τα περιλάβουμε όλα σε μια διαφάνεια. Αυτό που ήθελα να σας μεταφέρω ως μήνυμα είναι ότι ένα από τα πιλωτικά προγράμματα θα είναι η συζήτηση των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε στρατηγική σημασία χώρες για παράδειγμα ή σε χώρες με τις οποίες θα θέλαμε τέτοια συζήτηση για τις θεμελιώδεις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να είμαστε ε, υπερβολικά εξαντλητικοί, διεξοδικοί σε μία και μόνο διαφάνεια. Ε, Καταλαβαίνω τις αντιρρήσεις. Εδώ υπάρχουν αναφορές σε συγκεκριμένα, συγκεκριμένα θέματα τα οποία αποτελούν ένα κομμάτι των θεμάτων αυτών, ίσως όμως να είναι κάτι το οποίο διαφοροποιείται από το σύνολο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Καταλαβαίνω την παρέμβαση του κυρίου Σβέρ, υπάρχουν όμως κάποια παραδείγματα τα οποία αναφέρονται, ε, στα παραδείγματα αυτά υπάρχουν θεμελιώδη δικαιώματα, υπάρχουν όμως και κάποιες ε, προσπάθειες πρόληψης της παραβίασης, και αυτό θα μπορούσε να μην είναι συμβατό με τους βασικούς στόχους τους οποίους θέσατε αλλά με, ε, δευτερογενή επίπεδα προστασίας. Πάντως επαναλαμβάνω ότι η έρευνά σας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι ε, καλό θα είναι να προσπαθήσει κανείς να προωθήσει τη συζήτηση για τη νέα πολιτιστική διπλωματία. Αυτό το οποίο φέρνεται στην επιφάνεια και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε επανειλημμένα ζητήσει και στα πλαίσια του ψηφίσματος που μας υπενθυμίσατε, ότι οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνδέονται περισσότερο με αρμοδιότητες και αποστολές στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Εγώ σε λίγο θα έχω μία συνάντηση για τα θέματα της νέας σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τινησία. Θα συναντηθώ με κοινοβουλευτικούς από την Τινησία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της συνάντησης μία ώρα θα πρέπει να την αφιερώσουμε στα θέματα του πολιτισμού. Νομίζω ότι συμφωνούμε λοιπόν εδώ. Νομίζω ότι προϋποτίθεται η ύπαρξη ε, μιας σωστής δικτύωσης και γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι οι ενδείξεις και οι προτάσεις σας θα είναι πολύ χρήσιμες. Νομίζω ότι θα μπορέσετε να την παρουσιάσετε και σε άλλα φόρα και με την UNIC σαν παράδειγμα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και εύχομαι καλή δουλειά. Καλώς. Τελειώσαμε τη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ όλους, όλους τους συμμετέχοντες δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα κάτι. Α, ας ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγγνώμη. Δεν υποτιμώ σε καμία περίπτωση την παρουσία σας εδώ. Έχετε το λόγο. Δύο-τρία λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι σύντομος. Ήθελα ωστόσο να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαίρεται για την έκθεση που ακούσαμε. Τη μελέτη δηλαδή που έρχεται σε πολύ επίκαιρο χρονικό σημείο συνεργαζόμαστε με την, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων για την ανάπτυξη των πολιτιστικών δράσεων. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση που ακόμα συντάσσεται βέβαια, όμως ε, θα είναι σε ένα πλαίσιο people to people ε, βασισμένο στο νέο αυτό υπόδειγμα που ε, βασίζεται στην προπαρασκευαστική δράση την οποία συνενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προτείνουμε λοιπόν μια προσέγγιση εκ των κάτω, όπου δηλαδή τα πολιτιστικά ιδρύματα θα παίξουν ένα μείζωνα ρόλο. Ήθελα να τονίσω λοιπόν τη σημασία των σχέσεων που διαθέτουμε ήδη με τα πολιτιστικά ιδρύματα. Πρώτον, εκείνα είναι αυτά τα οποία ε, συνέταξαν την προπαρασκευαστική δράση μετά από σημαντικότατη διαβούλευση και στις χώρες μέλη και με τους στρατηγικούς εταίρους και με τις γειτονικές χώρες όχι μόνο λοιπόν με τα πολιτιστικά ιδρύματα αλλά και με τους ε, stakeholder εκ των κάτω όπως είπα από την βάση. Θα θυμάστε ίσως ότι και η Creative Europe χρηματοδοτεί ένα σχέδιο σε συνεργασία με το δίκτυο UNIC για να ενισχυθεί η στρατηγική ε, σκέψη και ε, η δημιουργία κλάστερ που θα είναι αυτών των ε, ομάδων δηλαδή ε, ιδρυμάτων που θα είναι οι φορείς οι οποίοι θα προωθήσουν τις ιδέες αυτές. Και βρισκόμαστε και στη διαδικασία έγκρισης μιας νέας στρατηγικής που θα ευθυγραμμίζεται και με αυτές που θα προτείνουμε. Και αυτό λοιπόν είναι πολύ καλοδεχόμενο στοιχείο. Τέλος δε, μέσα στα πλαίσια του εργαλείου εταιρικής σχέσης και του FBI ε, ξεκινούμε μια πλατφόρμα διπλωματίας που πάλι θα προωθηθεί από μια, μια σύμπραξη ε, πολιτιστικών ιδρυμάτων και θα δίνουν, θα παρέχουν συμβουλές στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά θα μας βοηθήσουν κιόλα στον σχεδιασμό και εκτέλεση δραστηριοτήτων ε, πολιτιστικής διπλωματίας αλλά και πολιτιστικής εκπαίδευσης. Τα πολιτικά ιδρύματα λοιπόν πάντοτε συμμετείχαν στο έργο μας και οι σχέσεις μας γίνονται όλο και πιο στενές. Ελπίζω δε ότι θα αποδειχθεί εξαιρετική συνεργασία μας μαζί τους και στο μέλλον. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ κύριε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις πληροφορίες που μας δώσατε από πλευρά της Γενικής σας Διεύθυνσης και της καινοτομίας εγώ υπολογίζω ιδιαίτερα και το είπα στον Επίτροπο χθε σε μια στενή συνεργασία για την νέα πολιτική της πολιτιστικής διπλωματίας με την κυρία Μογκερίνη και με τις διευθύνσεις ε, εκπαίδευσης πολιτισμού και καινοτομίας. και η ΕΟΝΙΚ μπορεί να πάρει μέρος στα πλαίσια αυτής της προετοιμασίας και έτσι θα ενισχύσουμε νομίζω την εξωτερική πολιτική διάσταση της Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Υπενθυμίζω σε όλους, κλείνοντας, ότι η επόμενη συνάντησή μας είναι στις 14 Μαρτίου και στις 15 Μαρτίου από τις 9 μέχρι τις 12.30 και από τις 3 μέχρι τις 6.30. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τη Γραμματεία, τη Γενική Διεύθυνση του Κοινοβουλίου και φυσικά ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Διευμηνία. Θα ήθελα να σας συζητήσω να βγείτε από την αίθουσα, θα συζητήσουμε με τους ε, συντονιστές παρακαλώ να βγείτε από την αίθουσα όσοι δεν παίρνετε μέρος στην επόμενη.